E Συνάδελφε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Επαναλαμβάνουμε τη σύνοδο. ανακοινώνω τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας για την εκλογή των αντιπροέδρων. Εψήφισαν 679, 16 άκυρα, 673 ε, ψήφισαν, 332 απόλυτη πλειοψηφία. Ε, οι υποψήφοι που πήραν την πλειοψηφία, την απόλυτη, και εκλέγονται είναι είναι η κυρία Κολάγια και ο κύριος Παπαδημούλης. Ο κύριος Κολάγια και ο κύριος Παπαδημούλης. Σε σχέση με τον κύριο Κολάγια, 426 ψήφοι και ο κύριος Παπαδημούλης 401. Ο κύριος Καστάλντο πήρε 284. Ο κύριος Κασοντεύσκη 261. Η κυρία Μπιτζότο 142. Συγχαίρω όσους εκλέγησαν. Βάσει του άρθρου 17, παραγραφός 2 του εσωτερικού κανονισμού, η ιεραρχία των Προέδρων βασίζεται στην σειρά με την οποία εξελέγησαν και ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν και την ε, ηλικία. Ε, παραμένουν ακόμα κάποιες έδρες όμως, μία έδρα συγκεκριμένα που πρέπει να καλυφθεί για την εκλογή των αντιπροέδρων λοιπόν. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά. Προτείνω λοιπόν στην Ολομέλεια Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Ωστόσο, πρέπει να ρωτήσω επισήμως και ρητός αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την πρόταση αυτή. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσεις. Θεωρώ ότι ισχύουν οι υποψηφιότητες όπως και στον προηγούμενο, το δεύτερο γύρο. Σωστά. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν παρεμβάσεις, οι υποψηφιότητες είναι αυτές του δεύτερου γύρου. Πρέπει όμως να σας ρωτήσω για σκοπούς διαφάνειας εάν όλοι οι βουλευτές στην αίθουσα έχουν μαζί τους την κάρτα τους. Υποθέτω ότι όλοι είστε σε θέση να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, συνάδελφε. Πρόεδρε, ακούσαμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα για κάποιες τεχνικές διευθετήσεις. Eh? Eh, Παρακαλώ, Πρόεδρε Τζάνι. Η ταυτότητα και η δημοκρατία επιμένει να ψηφίσουμε όπως και στους προηγούμενους γύρους με κανονικά ψηφοδέλτια. Άρα, η πρόταση για ηλεκτρονική ψηφοφορία, να την ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε την πρόταση αυτή καθεαυτή. C'è qualcuno che si esprime a favore Υπέρ της ηλεκτρονικής με δηλώσει, με δηλώσει πρέπει, όχι με ανάταση χειρό. Κάποιο πρέπει να υπερασπιστεί την πρόταση. Θέλει κάποιο να λάβει το λόγο. Ο κύριος Κόρμπετ. Yes, Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα κερδίσουμε και χρόνο με τη χρήση του συστήματο ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το σύστημα υπάρχει, το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει, λειτουργεί τέλεια, εξακολουθεί να ε, εξασφαλίζει μυστική ψηφοφορία και μας επιτρέπει να είμαστε ταχύρυθμοι και αποτελεσματικοί. Allora, mettiamo in votazione la proposta del voto. Οπότε, ψηφίζουμε για την διαδικασία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όσοι είστε υπέρ, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σα. Κατά. Αποχές. Ωραία. Γίνεται δεκτή η πρόταση. Però per rispondere alla Όμως, για να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση για το δεκάλεπτο διάλειμμα, ας κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών και μετά ευθύ αμέσω ψηφίζουμε.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 No, is el No, No, no, no, no, no. Allora, colleghe, e colleghi. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καθίστε παρακαλώ.